Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Ξεκινήσαμε χθες. Ε, προέδρευε ο κύριος Σάβαρμα, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που με αντικατέστησε. Καταλαβαίνετε ότι εχθές ήταν η επομένη του πρώτου γύρου των εκλογών ε, που ε, αφορά και την Ευρώπη στη Γαλλία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την κατανόηση και ευχαριστώ και τον κύριο Σάβαρμα. Ε, έγινε η συνεδρίαση των συντονιστών σήμερα το πρωί στις 9.30 και θα ήθελα να σας πω ότι αποφασίστηκε ο διορισμό των εισηγητών για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Επιβεβαιώνουμε την έκθεση και ο εισηγητή θα είναι ο κύριο Όλμπρεχτ και η κυρία Τομά. Ε, μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων, Λεβαντόφσκι και Ντεπρέ επιβεβαιώνονται. Και επίσης ε, καταλήξαμε στη σύσταση μιας ομάδας εργασίας για τα εσωτερικά θέματα, για την κατάρτιση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ομάδα του Κοινοβουλίου θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους ε, του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών και δημοκρατών και οι άλλες πολιτικές ομάδες θα έχουν από έναν εκπρόσωπο. Ε, βεβαίως ε, θέλουμε όσοι ήταν οι εισηγητές από την έναρξη της θητείας να είναι τα μέλη τα οποία θα ορίσει η ομάδα τους και φυσικά οι πολιτικές ομάδες γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τους αντιπροσωπεύσουν και θα μας τα κοινοποιήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σάρβαμα για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Μετά από έτσι που επέβαλε η Φιλανδία, ε, Νότια Network System. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ λοιπόν και πάλι δυστυχώς πρέπει να συζητήσουμε για τρίτη φορά μία αίτηση για θέματα πληροφορικής από τη Φιλανδία. Είναι το 1 πέμπτο όλων των αιτήσεων ε, στο τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Ε, Είχαμε 15 μέχρι τώρα για το Ταμείο, για το ICT και αυτή είναι η τρίτη από τη Φιλανδία. Η οποία βέβαια είναι κολοσσός ε, σε θέματα τεχνολογίας και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Η Nokia Network Systems απέλησε 945 άτομα και οι 821 από αυτούς είναι δικαιούχοι του Ταμείου, είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι. Και φυσικά το Ταμείο προσαρμογή ε, στην Παγκοσμιοποίηση θα καλύψει ω συνήθω το 60% του κόστους, 2,6 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, των συνολικών 4,2 εκατομμυρίων. Τι κάνω στη Φιλανδία Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης ε, συνεδριάζει με εκπροσώπους των ενδιαφερομένων και των εργαζομένων σε αυτή την περίπτωση και καταρτίζουν ε, ένα πακέτο ε, εξατομικευμένες υπηρεσίες και είναι προς το συμφέρον το δικό μας ε, για τα θέματα ελέγχου του προπολογισμού να δούμε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Και σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της αίτηση της Φιλανδίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ε, μετεκπαίδευση για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων για τους εργαζομένους, διότι ε, είναι τσοκαριστικά τα στατιστικά στοιχεία. Το 21% των απολυμένων σε αυτή την περίπτωση, των, από αυτούς τους 945 ανθρώπους, ήταν άνω των 55 ετών, το 21%. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να μπορέσουν να βρουν μια νέα θέση εργασίας και Εκεί ακριβώς θα θέλαμε να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του Ταμείου και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δίνεται λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και τα υπόλοιπα χρήματα πηγαίνουν σε αρκετά πράγματα, ε, ρυθμιστικά μέτρα, ε, υπηρεσίες επιχειρήσεων κλπ. Και επίσης ε, το δίκτυο EURES ε, χρησιμοποιείται στη Φιλανδία για ε, τα θέματα αυτά. Τα μέτρα λοιπόν εξέβρεση νέων θέσεων απασχόληση ξεκίνησαν να εφαρμόζονται πριν καν υπάρξει χρηματοδότηση από το Ταμείο Προσαρμογή και την απόφαση τη Ένωση και τα, η Φιλανδία ε, μας έδωσε όλες τις πληροφορίε ε, για την αίτηση χωρίς καμία καθυστέρηση. Ε, πρόκειται για κάτι λοιπόν το οποίο θα προχωρήσει ο, ομαλά κατά την άποψή μας. Η Επιτροπή Έμπλου θα γνωμοδοτήσει βεβαίως και αυτή τη φορά ακούμε και κάποιες φήμες ότι μπορεί να υπάρξει και κάτι ασυνήθιστο, κυρίως ε, δεδομένου ότι ε, Συνήθως αυτά είναι πράγματα ρουτίνας. Θα δούμε σε τι θα καταλήξει η Επιτροπή Απασχόλησης. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 28 Απριλίου, την Παρασκευή δηλαδή, σε τρεις μέρες, στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σάβερμα. Η κυρία Γιατενμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα μιλήσω φιλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Για να γίνω πιο κατανοητή. Είναι η τρίτη φορά που εξετάζουμε μια αίτηση του τομέα της πληροφορικής από τη Φιλανδία. Όπως ε, είπε ο κύριος είναι μια δυσάρεστη θέση. Θα προτιμούσα να μην βρίσκομαι δηλαδή σε αυτή τη θέση, αλλά έχουμε αυτή την αίτηση που έχει κατατεθεί, πληρεί τα κριτήρια και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τη στήριξη. Η κατάρρευση της Νόκια ε, ήταν η μεγαλύτερη επιχειρηματική τραγωδία στη Φιλανδία και έχει επηρεάσει χιλιάδες ανθρώπους στη Φιλανδία και εξακολουθεί να πλήττει ε, εργαζομένους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει συσταθεί ακριβώς για να βοηθήσει όσους ε, χάνουν τη δουλειά τους ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης και της ε, παγκόσμιας κρίσης. Για να βοηθήσουμε τους ανέργους να βρουν και πάλι δουλειά και έτσι αυτοί οι υπάλληλοι της Νόκια χρειάζονται τώρα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να βρουν νέες θέσεις απασχόλησης. Και αυτός είναι ο σκοπός του Ταμείου. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει εδώ ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο χρήζει προσοχή. Η ανακύκλωση ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά αυτόν τον τρόπο είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από αυτό το Ταμείο και πιο συγκεκριμένα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι όντως αποκτούν νέες δεξιότητες και κατά πόσο αυτές οι νέες δεξιότητες αποκτώνται χάρη στο καινούριο ταμείο ή μήπως θα μπορούσαν να αποκτηθούν με άλλους τρόπους. Παρ' όλα αυτά, η αίτηση αυτή πληρεί τα κριτήρια και εγώ στηρίζω να ε, υπάρξει στήριξη από το Ταμείο. Βεβαίω το σημειώνουμε. Δεν έχει στήσει κανείς άλλο τον λόγο. Ένα αυτό το Ταμείο μπορεί να αξιοποιηθεί πριν από την απόλυση, ούτω ώστε δηλαδή η επιχείρηση να προσαρμοστεί στην παγκοσμιοποίηση, αυτό θα ήταν μια πρόοδο. Γιατί εδώ πρώτα περιμένουμε να υπάρξουν απολύσεις και μετά παρεμβαίνουμε. Τέλος πάντων. Ο κ. Σαββάρμα μας είπε ότι οι τροπολογίε πρέπει να κατευθούν μέχρι τις 28 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. Στην Επιτροπή Προλογισμού θα ψηφίσουμε στις 11 Μαΐου και στην Ολομέλεια στις 16. Στις 27 Μαρτίου η Επιτροπή μας υιοθέτησε δύο εκθέσεις σχετικά με την ε, εντολή της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μπήκαμε λοιπόν τώρα στην φάση των τριμερών διαλόγων. Η Επιτροπή μας αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ξεκινήσει πραγματεύσεις επί αυτή τη βάση, αυτής της ψηφορίας δηλαδή βάση του άρθρου 69 παραγράφου 3 του στον κανονισμού. Μετά από κάθε τεμερή διάλογο θα πρέπει να υπάρξει μια σύνοψη εξ ονόματος της ομάδας διαπραγματεύση κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίας της Αρμόδιας Επιτροπής. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε τώρα τους Φρίντε Μουρισάν και Ζαμπάρ για να ακούσουμε ακριβώς τι συνέβη στο τελευταίο τριμερή διάλογο στις 12 Απριλίου. Παρακαλώ κυρία Γκαρδιά Θεμπάλ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο αντιπρόεδρος ο κύριος Μωρεσάν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Θα σας κάνω εγώ λοιπόν τον απολαγισμό της συνεδρίασης στις 12 Απριλίου, αμέσως πριν τις ε, διακοπές της Μεγάλης Εβδομάδας. Ε, Νομίζω ότι ήταν αρκετά καρποφόρα η συζήτηση, ε, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που συναντούσαμε τη Μαλτέζικη Προεδρία για να συζητήσουμε την έκθεση για την εξωτερική εντολή της ε, Τράπεζας Επενδύσεων και ε, καθορίσαμε δέκα σημεία στα οποία θέλαμε να κάνουμε μια πιο γενική και πολιτική συζήτηση για να καταλήξουμε σε κάποιες θέσεις και μετά στον επόμενο τριμερή διάλογο θα κάνουμε συζήτηση κατάρθρο. Αυτά τα δέκα θέματα Τα κατηγοριοποίησαμε, αποφασίσαμε ότι τέσσερα εξ αυτών μπορούν να συζητηθούν ήδη σε τεχνικό επίπεδο γιατί σε πολιτικό επίπεδο συμφωνούμε οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ένταξή τους, όλα όσα έχουν να κάνουν με την πολιτική της ισότητας. Ο νέος ε, στόχος ε, που προστίθεται αυτός ο τέταρτος νέος στόχος της εξωτερικής ε, εντολής της ε, Τράπεζης Επενδύσεων ε, για τους πρόσφυγες και το θέμα της διαφάνειας και της υποβολής εκθέσεων. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι στα τέσσερα αυτά θέματα, δεδομένου ότι υπάρχει συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο, μπορούμε να τα συζητήσουμε σε τεχνικό επίπεδο. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες της τεχνικής ομάδος, αν και ορισμένες φορές θεωρούμε όντως ότι ολοκληρώθηκε η πολιτική συζήτηση και πρέπει να συμφωνήσουμε επί της διατύπωσης και να ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε τις εργασίες. Ορισμένες φορές, ε, ε, ο, όπως βλέπουμε και στο θέμα της διαφάνειας και της υποβολής εκθέσεων, υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσον πρόκειται απλώ για τεχνικό θέμα και ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε και πάλι σε πολιτικό επίπεδο. Κατόπιν έγινε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος ε, και τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ένας από τους στόχους πρέπει να είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει ακριβώς στο πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ποιες δράσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τι θα πρέπει να ενισχύσουμε. Από το Συμβούλιο μας έλεγαν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι δεν αναφερόμαστε σε ενισχύσεις αλλά σε έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα και επομένω αυτό δυσχεραίνει λίγο τα πράγματα. Εμείς επιμείναμε ότι πρόκειται για προτεραιότητα και ότι ένας από τους λόγους της μετανάστευσης είναι προφανώς και η κλιματική αλλαγή και επομένω δεν ε, θα ε, εγκαταλείψουμε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη χρηματοδότηση έργων προς αυτή την κατεύθυνση σε καμία περίπτωση. Το Κοινοβούλιο ε, θα εμείνει σε αυτό το ζήτημα. Ε, αναφερθήκαμε επίσης και στην ευελιξία που είναι μία από τις ανησυχίες του Συμβουλίου στο σημείο αυτό τους είπαμε ότι στο Κοινοβούλιο, επειδή δεν υπήρχε τροπολογία του Κοινοβουλίου, δεν υπήρξε χρόνο να συζητήσουμε ει βάθος και είναι και κάτι το οποίο θα συζητήσουμε άλλωστε στην επόμενη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών και φυσικά υπάρχουν και τα πιο ακαθόδη ζητήματα, επί των οποίων σίγουρα θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά στου επόμενου μήνε. είναι τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη φορολόγηση, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, τις ε, ε, χώρες που δεν ε, συνεργάζονται και την επιθετική φορολογική πολιτική. Σε γενικές γραμμές, ναι, μεν τα τρία θεσμικά όργανα είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως διαφωνίες για τα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Και υπάρχουν και αρκετές αποκλήσεις σε νομικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι μπορούμε να βάλουμε νομικό σε ένα κομμάτι χαρτί και ε, πιστεύουμε ότι τρεις νομικές υπηρεσίες των ε, θεσμικών οργάνων θα πρέπει να ξεκινήσουν να συνεργάζονται και να γίνει μια συζήτηση ε, για το τι θα ήταν ενδιαφέρον και τι ε, μας επιτρέπεται από νομική σκοπιά να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη συμφωνία. Σε αυτό το θέμα της φορολόγησης προκύπτει και ένα πρόβλημα επιπλέον διότι είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε στους επόμενους μήνες σε τρεις παράλληλες εκθέσεις. Σε αυτήν για την εξωτερική εντολή του ε, Ταμείου Επενδύσεων, στο Ταμείο Εξωτερικών Επενδύσεων, το οποίο εγκρίναμε χθε και αύριο θα δοθεί και το πράσινο φως να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και το σχέδιο Juncker. Επομένως θα ήταν ενδιαφέρον να βρούμε έναν τρόπο να συντονίσουμε τις διαπραγματεύσεις σε αυτές τις τρεις εκθέσεις για το θέμα αυτό. Αλλά αυτό βεβαίως συζητήθηκε ακροθυγώς λίγο στον τριμερή διάλογο ότι αφορά και τρεις διαφορετικές εκθέσεις και καλό θα ήταν να γίνει μία διαπραγμάτευση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις τρεις εκθέσεις αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ ε, αρχικό στάδιο. Μετά έγινε η συζήτηση για το ποιο ε, θα είναι ο υπεύθυνος της διαχείριση του Ταμείου. Εδώ και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η διαχείριση αυτού του Ταμείου, ε, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στοιχείων ενεργητικού, αλλά ε, η ε, Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν θέλαμε να συνεχίσουμε περισσότερο, ζητήσαμε να γίνει μια προσπάθεια. Θεωρούμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον η διαχείριση του Ταμείου να διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε ε, να κάνουμε αυτό το οποίο προτείνει για το μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει ενιαία διαχείριση όλων των ταμείων εγγύησεων και προς το παρόν δεν υπήρξε περαιτέρω πρόεδρος και βεβαίως το πιο σύνθετο ζήτημα, στο οποίο ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία στο μέλλον, έχει να κάνει με τα ανώτατα όρια και την ε, περιφερειακή κατανομή. Δεν το συζητήσαμε καν το θέμα της περιφερειακής κανονομής, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το, ε, και να συμφωνήσουμε το συνολικό ποσό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική εντολή ε, σίγουρα και επίσης να υπάρχουν και κάποια προφανή στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να διευρύνουμε το ανώτατο όριο της εξωτερικής δανειοδότησης της Τράπεζας Επενδύσεων και θεωρούμε ότι είναι λίγα χρήματα για όλα όσα μπορούν να γίνουν. Και με μια πολύ μικρή επιπλέον προσπάθεια στον προπολογισμό θα μπορούσαμε να αυξήσουμε πάρα πολύ τις επενδύσεις στις χώρες ε, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εξωτερική εντολή της Τράπεζας Επενδύσεων. Επομένως, ε, εξακολουθούμε να πιέζουμε και να απαιτούμε από το Συμβούλιο να ε, ε, εξετάσει δυνατότητες να αυξήσουμε τα ανώτατα όρια της εξωτερικής εντολής και κυρίως ε, τους υπενθυμίσαμε να λάβουμε υπόψη ότι τουλάχιστον εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε την αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου που σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παγκόσμιο αποθεματικό για τις ε, δεσμεύσεις για να τα χρησιμοποιήσουμε πλέον και για τη μετανάστευση και όχι μόνο για την απασχόληση, άρα έχουμε μια επιπλέον δυνατότητα. Με αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Δεν ε, συζητήσαμε τα θέματα κατάρθρων, γιατί θεωρούμε ότι για πρώτη επαφή έγιναν αρκετές ε, ανταλλαγές απόψεων και επικεντρωθήκαμε και σε αρκετά σημαντικά θέματα. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει την Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε και συνεδρία των σκιωδών πριν από τον τριμερή διάλογο, στην οποία θα συζητήσουμε κάποια από αυτά τα θέματα και θα ξεκινήσουμε και τη συζήτηση κατάρθρων, ε, βλέποντας τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ε, οριστικοποιημένο και θέσεις του Κοινοβουλίου και κάποιες θέσεις του Συμβουλίου και θα δούμε και ποια θέματα θα πρέπει να συζητήσουμε στον επόμενο τριμερή διάλογο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Έντερ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Για να ευχαριστήσει την ΕΝΤΕΡ για την δουλειά που έχει κάνει. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να έρθει ο Σικφρίντ Μερισάν για να ξεκινήσουμε την ομάδα παρακολούθησης. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Ξέρω ότι είναι καθοδόν ο Σίκφριντ. Έρχεται λοιπόν. Donc la séance est suspendue quelques minutes. Ένα διάλειμμα ορισμένων λεπτών λοιπόν.